Eh, Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε την συνεδρίαση την απογευματινή. Καταρχάς, έχουμε το θέμα άστο της ημέρας που είναι η παρουσίαση του πακέτου μεταρρυθμίσεων από πλευρά της Επιτρόπου της κυρίας Δαμανάκη που ε, ε, έχει εγκριθεί επιτέλους αυτό το πακέτο και καλή στιγμή μάλιστα εγκρίθηκε. Και μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε παραπέρα. Παρόλο που είναι διαθέσιμο μόνο σε τρει γλώσσε το κείμενο, καλώ ήρθατε λοιπόν κυρία Επίτροπε. Θα σα δώσω το λόγο, ούτω ώστε να μπορέσετε να μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι, είναι η πρώτη φορά που ένα επίτροπος ομιλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την μεταρρύθμιση τη κοινή αληθική πολιτική σαν ισότιμος υποχρεωτικό εταίρος του Συμβουλίου, του Κοινοβούλιο. Σήμερα είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και αν συνεργαστούμε, σήμερα θα είναι η απαρχή ε, μιας ιστορικής αλλαγής. Γνωρίζουμε όλη την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Έχουμε μείωση αποθεμάτων κάτι που σχετίζεται με την υπεραλίευση και την απόρριψη, σχετίζεται με το πολύ μεγάλο δυναμικό, υπερβολικό δυναμικό των σκαφών και συνδέεται με τις επιδοτήσεις. Το κεντρικό μας σύστημα μας καταδικάζει σε μικροδιαχείριση που είναι κάτι δαπανηρό για τον φορολογούμενο. Έχουμε μελέτες που αποδεικνύουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 75% των αποθεμάτων είναι αντικείμενο υπεραλίευσης. Ρίξτε μια ματιά σε αυτή τη διαφάνεια, ελπίζω να είναι σωστή που δείχνει ότι οι αλληλείς μας όλοι αλλιεύουν ένα κλάσμα αυτού που αλλίευαν τη δεκαετία του 90. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα για τον αλληλευτικό μας τομέα ε, που δεν είναι επικερδής. Να σας δείξω πώς εξελίχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες οι στόλοι μας. Η πάνω γαλάζια γραμμή δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε λιγότερα σκάφη κάθε χρόνο, ακόμα έχουμε μία αύξηση του 3% όσον αφορά το δυναμικό του στόλου. Γιατί, διότι εξυγχρονίσαμε τα σκάφη μας και φυγήσαμε καινούρια και αυτά είναι πολύ πιο προδευμένα τεχνολογικώς. Έτσι τα τελευταία χρόνια έχουμε εξυγχρονισμό που κινείται παράλληλα με την αύξηση του δυναμικού. Και τώρα κοιτάξτε τα πραγματικά καταστροφικά μαντάτα, κυρίως ότι αυξήθηκε το δυναμικό παρά τα τεράστια ποσά χρημάτων των φορολογωμένων που ε, δόθηκαν για, τον, για την καταστροφή των πλοίων, για τον αφοπλισμό τους, πάνω από 906 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ανάμεσα στο 2006 και 2006 και μόνο. Και είχαμε σχεδόν μηδέν αποτέλεσμα παρόλες τις δαπάνες. Γι' αυτό πρόσφατα λάβαμε και μια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου περί των δαπανών αυτών και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη για τον επόμενο χρόνο. Λοιπόν, τι θα συμβεί αν δεν σπάσουμε αυτό τον φαύλο κύκλο. Λοιπόν, να σας πω. Σύμφωνα με την αξιολόγηση συνεπιών που κάναμε, αν δεν γίνει μεταρρύθμιση, μόνο 8 αποθέματα από τα 136 θα είναι σε επίπεδο βιώσιμο το 2022. Με άλλα λόγια, θα χάσουμε ένα αλλιευτικό απόθεμα μετά το άλλο διαδοχικά με ενδεχόμενη λεσιδωτή αντίδραση για το οικοσύστημα που είναι κάτι δύσκολο να προβλεφτεί. Ποιο θα είναι. Τι γίνεται με τη βιομηχανία μας. Θα αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερη οικονομική πίεση ο τομέας αυτός. Τα στοιχεία εδώ δείχνουν ότι σήμερα το 35% των επιχειρήσεων ε, λειτουργούν με απώλειες. Με την ισχύουσα πολιτική. 35% των επιχειρήσεων ε, λειτουργούν με απώλειες. Εάν δεν κινηθούμε θα χάσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην αλληλεία, μεταποίηση, μεταφορές, υποδομές λιμένων και λιανεμπόριο. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στις παράκτιες περιφέρειές μας, των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται από την αλληλεία. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα η αλληλεία μπορεί να συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού σε τρόφιμα και σε οικονομική ανάπτυξη. Μπορεί και να διοχετευτεί και πρέπει να διοχετευτεί η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 και να γίνει αλληλεία πηγή πλούτου για του αλληλεί και για τι παράκτιε κοινότητε. Για να το πετύχουμε αυτό, η μεταρρύθμιση έχει τρει πυλώνε: βιωσιμότητα, αποδοτικότητα και συνοχή. Ας αναφερθώ στο πρώτο πυλώνα, βιωσιμότητα, περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική βιωσιμότητα. Είναι στην καρδιά αυτού του πακέτου και εκεί περιέχονται διάφορα στοιχεία. Πρώτα, θέλουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Αυτή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση θα πρέπει να γίνει μια νομική υποχρέωση. Αυτό συμφωνήθηκε στο Johannesburg το 2002 και είναι και ένα κομμάτι του UNCLOS, δεν αφορά μόνο τη συνθήκη του Johannesburg, αλλά επίσης και ένα τμήμα του UNCLOS και των διεθνών υποχρέωσεών μας. Τα απορίσματα της Παγκοσμίου Τραπέζης όσον αφορά τα βυθισμένα δισεκατομμύρια, η σχετική μελέτη, την οποία παραλάβαμε, λέγεται Sunken Billions, τα βυθισμένα δισεκατομμύρια. Ε, και τα αποτελέσματα τη εξοργή συνεπειών είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα, ηλίου φαϊνότερα. Εάν ανοικοδομήσουμε, αν αποκαταστήσουμε τα λεφτικά αποθέματα, μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλα επιπλέον 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ ε, για την λεφτική βιομηχανία μας σε μια δεκαετία. Αν επιτρέψουμε την ανάκαμψη των αποθεμάτων, δεν πρόκειται να έχουμε προβλήματα για τον τομέα μας, όπως λέγουν πολλοί. Ε, έχουμε πολύ καλή αξιολόγηση συνεπιών, ακριβέστατη, που αποδεικνύει ότι αν καταφέρουμε χειριστούμε σωστά ε, στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση τα αποθέματα, θα έχουμε προστιθέμενη αξία για τη βιομηχανία μας ύψους 2,7 δις για μία δεκαετία. Βλέπετε σε αυτή τη γραφική παράσταση παραδείγματα για την επίτευξη του μέγιστου ε, βιωσίμου επίπεδου ε, απόδοσης και πώς μπορεί να φαίνεται η καμπύλη των αποθεμάτων. Βλέπετε εδώ το παράδειγμα ε, του Βακαλάου στο Βόρεια Αρκτική και στη Βόρεια Θάλασσα επίσης και βλέπετε πώς τα αποθέματα ανακάμπτουν και βελτιώνονται και πώς μπορούν να επέλθουν και πρόσθετα κέρδη για την βιομηχανία. Ένα άλλο στοιχείο για τη βιωσιμότητα θα πρέπει να σταματήσουμε τις απορρίψεις, διότι το να πετάμε τα τρόφιμα σε έναν πεινασμένο κόσμο είναι κάτι που καταστρέφει την εικόνα μας και υπονομεύει τη συλλογή στοιχείων. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς ποια είναι τα αλλιεύματα, η ποσότητα των αλλιευμάτων. Γι' αυτό προτείνω να έχουμε βέβαια μια μεταβατική περίοδο, αυτό περιέχεται στην πρότασή μας, αλλά στο τέλος θα πρέπει να εκφορτώνονται όλα τα αλλιεύματα και να μετρώνται και να λαμβάνονται υπόψη στις ποσοστώσεις και να συγκρίνονται. Θα πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο λήψης αποφάσεων και αυτό δίνει τροφή στο δεύτερο πυλώνα του, ε, της πρότασής μας, την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα. Τη χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε νέα μορφή διακυβέρνησης. Να είναι καλής αποτελεσματικός σημαίνει ότι αφήνει τις πολιτικές αποφάσεις για το πολιτικό επίπεδο, δηλαδή Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Και οι τεχνικές αποφάσεις όσον αφορά τα μάτια των δικτυών, περιορισμούς για τα, για τα εργαλεία που χρησιμοποιεί την αλληλεία, το αφήνουμε στα κάτι μέλη και στην αλληλευτική βιομηχανία. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Γι' αυτό σα προτείνω εσεί και το Συμβούλιο να θετήσετε παραδείγματο χάρη μακροπρόθεσμο σχέδιο για το γάδο το Ατλαντικό. Α το πάρουμε αυτό σαν παράδειγμα. Για το Μερλούκιο, συγγνώμη θα πρέπει ο μελούκιος να μείνει πάνω από τα επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Όλα τα κάτι μελη εκεί που έχουν ε, τα σκάφη που αλλιεύουν για το μερλούκιο θα πρέπει να συμφωνήσουν τι μέτρα θέλουν. Παραδείγματο χάρη θα πρέπει να περιγράφουν συγκεκριμένο υλικό που χρησιμοποιείται περιορισμένο αριθμό ημερών στη θάλασσα ή να κλείνει η να κλεινει η αλλιεια για δύο μήνε. Ε, εκεί θα αποφασίσουμε για όλα αυτά τα μέτρα. Δεν μας νοιάζει ποια μέτρα θα επιλεγούν από αυτούς. Μπορούν να επιλέξουν τα δικά τους. Εδώ μιλάμε για περιφερειοποίηση. Αυτό που μετρά για μας πώς θα πετύχουν, ότι θα πετύχουν τους στόχους. Όχι πώς, ότι θα πετύχουν τους στόχους. Μπορεί να πετύχουν τους στόχους με το δικό τους τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ο φάρος, αν θέλετε, που θα φωτίζει το δρόμο. Αυτό που θα θέλαμε θα ήταν να δείχνουμε την πορεία. Τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες και η βιομηχανία θα πρέπει να είναι στο πιδάλιο του σκάφους και να φύγουν τα βράχια βέβαια. Το θεωρώ ότι είναι τεράστιο όφελος αυτό για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες, διότι γίνονται ιδιοκτήτες των μέτρων, υπάρχει λιγότερη μικροδιαχείριση από πλευράς Βρυξελών, διότι μπορούν να θεσπίσουν μέτρα μαζί με τον τομέα. Αυτό είναι σημαντικό, διότι να εκμεταλλευτούμε πλήρως την τεχνογνωσία τους. Τι γίνεται λοιπόν με τι οργανώσει των παραγωγών. Με αυτή τη μεταρρύθμιση, οι οργανώσει των παραγωγών θα έχουν ένα πραγματικό ρόλο όσον αφορά τη διαχείριση των αλευτικών αποθεμάτων. Μπορούν παραδείγματο χάρη να εξασφαλίσουν ότι τα μέλη δεν ξεπερνούν τι ποσοστώσει. Μπορούν να εθετήσουν πιο επιλεγμένο υλικό και εργαλεία που χρησιμοποιούν την ελεία και μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη του αφορά τη σημασία που έχει το να λιεύει κανεί υπεύθυνα. Μια περιφερειοποιημένη πολιτική, όπω σα προανέφερα και περιέγραψα, είναι απλούστερη στην εφαρμογή τη και φθηνότερη για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Θέλουμε επίση να πετύχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εμπασματικότητα εισάγοντα μεταφερόμενε ε, εκχωρήσει, αδειοδοτήσει για την αλεία. Εδώ τουλάχιστον προσπαθούμε με ένα σπάρο να σκοτώσουμε δύο τριγώνια. Διότι θα μειωθεί ο στόλος και θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την απαγόρευση της απόρριψη. σε έναν αριθμό χωρών που ήδη χρησιμοποιούν τα μεταφορόμενε αυτέ αληφτικέ άδειε, εκχωρήσει. Ε, μειώθηκε ο στόλος πολύ περισσότερο παρά με, διάφορα, με πολλά χρήματα που έχουν διατεθεί στην ε, Δανία. Ο, ο στόλος έχει μειωθεί κατά 30% παράκτιος και το πελαγικός ε, κατά 50%. Ο βένθο πελαγικός μάλλον κατά 30% και ο πελαγικός κατά 50%. Λοιπόν, ήδη εξάσατε κάποιες αμφιβολίες για αυτά τα προβλήματα. Οπότε έλαβα υπόψη αυτά που είπατε και προτείνω συγκεκριμένες ρήτρε διαφύλαξης, μέτρα προφύλαξης. Πρώτα απ' όλα οι μεταφορές περιορίζονται στο εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, μόνο οι αλληλείς μπορούν να αγοράσουν αυτές τις άδειες αλευτικές, τα δικαιώματα αυτά. Μόνο οι διοκτήτες των σκαφών, όχι πάντες. Τρίτον, τα κράτη-μέλη μπορούν να εξαιρέσουν ε, στόλου μικρή κλίμακα στο σύστημα, έτσι ε, περαιτέρω τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν πρόσθετα μέτρα διαφύλαξη να αποφύγουν υπερβολική συγκέντρωση και αν το θέλουν αυτό και να εξασφαλίσουν ένα, μια οικονομική απόδοση, οικονομικό συσχετισμό. Αλλά αυτέ οι άδειε δεν θα εξορθολογήσουν μόνο του τόλου, αλλά θα βοηθήσουν να σταματήσουν και απορρίψει. Πώ θα γίνει αυτό. Στο μέλλον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες σκαφών να αλλάζουν τις χωρίς αδειοδοτήσεις μεταξύ τους, να τις μισθώνουν, να τις πολλούν. Αυτό θα επιτρέψει Αλληλής να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτα μπορούν να αποκτήσουν ένα συνδυασμό ποσοστώσεων σύμφωνα με το μέτρο τους, με τις ανάγκες τους και τον τρόπο που αλλιεύουν και δεύτερον, όταν ένα καπετάνιο θεωρεί ότι δεν έχει ποσοστώσει για το 30% του ελίευματός του, τότε μπορεί να στείλει σήμα στην ε, οργάνωση παραγωγών σε πραγματικό χρόνο, ούτω ώστε να ανιστώσει αρκετή ποσόστοση. Έτσι θα αποφύγουμε ε, τις απορρίψεις. Οπότε έρχομαι στην κοινωνική πλευρά της ε, διότι αυτή η μεταφορά των αδειών ε, ε, ε, Αλλιέ θα δώσει οικονομική ασφάλεια σε αυτού που θέλουν να ζήσουν από τον τομέα. Και επειδή ένα επικερδής αλληλευτικός τομέας θα δώσει στους αλληλείς και στους οικογένειε του οικονομική ασφάλεια. Άρα θα δώσει και ασφαλή ανάπτυξη και προοπτικές στις παράκτε κοινότητες οι οποίες κοινότητες αυτές, οι παράκτες είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την ε, Ευρώπη. Και τώρα ερχόμαστε στον τρίτο πυλώνα, συνοχή όλα τα τμήματα της πολιτικής από τις οργανώσεις και την οργάνωση αγοράς, υδατοκαλλιέργεια, εξωτερική διάσταση μέχρι οικονομική υποστήριξη θα πρέπει να υποστηρίζουν την βιωσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Συνοχή τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όσο οι καταναλωτέ θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι αγοράζουμε, εμεί οι καταναλωτέ θα ξέρουμε τι έχουμε δικαίωμα να αγοράσουμε. Άρα βελτιώνεται και το του ώστε να δίνονται επακριβεί πληροφορίε όσον αφορά την πρόλευση του προϊόντο και τον τρόπο παραγωγή αυτού. Επειδή παράλληλα καταπολεμούμε και την παράνομη αλληλεία και δημιουργούμε μια νοοτροπία συμμόρφωσης, οι καταναλωτέ θα γνωρίζουν ότι αυτό που αγόρασαν ε, αλλιεύτηκε με βιώσιμο τρόπο. Είτε το αγοράζουν για τους δικούς μας αλληλείς από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν αγοράζουν το προϊόν ως εισαγόμενο προϊόν. Αλλά η συνοχή για μένα επίσης σημαίνει το να παραδεχόμαστε ότι αυξάνεται η ζήτηση για τα ψάρια και δεν μπορεί αυτό να καλυφθεί μόνο από την αλία. Γι' αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε καλύτερα τις ιδετοκαλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια πραγματική αλλαγή εδώ, όχι μόνο για να διευρύνουν τον τομέα, αλλά πραγματική αλλαγή. Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να φέρει ανάπτυξη έξυπνη και καινοτόμα και στις περιοχές παράκτης αλλά και τις εσωτερικές των χωρών. Και γι' αυτό σημαντική ε, δραστηριότητα έχει θέσει στο βασικό κανονισμό. Θα βοηθήσει και ανάπτυξη και τη ενδοχώρα. Θα δώσει στρατηγικέ κατευθύνσει γραμμέ σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για τι διδοκαλλιέργειε με κοινέ προτεραιότητε και στόχου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει τότε να θεσπίσουν πολιετή σχέδια για να αναπτύξουν τη βιομηχανία αυτή, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και να προσφέρουν στους εμπορευόμενους μια δίκαιη πρόσβαση σε χώρο και σε ύδατα. Συνοχή επίση σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε εξίσου βιώσιμοι στη δική μας εξωτερική πολιτική όπως είμαστε και στα δικά μας ύδατα. Γι' αυτό προτείνω βιώσιμες αλληλευτικές συμφωνίες. Μια νέα γενιά συμφωνιών που θα επικεντρώνονται επί των ιδίων αρχών που εφαρμόζουμε στο εσωτερικό. Η Ένωση θα πρέπει να συνάπτει μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα μόνο αν υπάρχει πλεόνασμα από που δεν χρησιμοποιείται από τον τόπιο τομέα και αν η επιστήμη μας λέει ότι είναι ασφαλές να αλληλευθούν αυτά τα αποθέματα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών θα αποτελεί ένα τμήμα αναπόσπαστο κάθε συμφωνίας. Τέλος, ας πω μερικά λόγια για την χρηματοδότηση. Κυρίες και κύριοι, είναι αυτή είναι δύσκολη οικονομική καιρή πολέμησα για ένα επαρκέ επίπεδο χρηματοδότηση με του συναδέλφου μου του επιτρόπους και η λογική είναι απλή. Να εξασφαλίσουμε την επιτυχία τη μεταρρύθμισης. Για το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε προπολογισμό που μοιάζει με τον ισχύοντα. Θέλω να το χρησιμοποιήσω τον προπολογισμό αυτό για να προωθήσω την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και ευφυή και ενταξιακή ανάπτυξη στι παράκτιε περιοχέ. Αργότερα, το τρέχον έτος, θα παρουσιάσω το δημοσιονομικό κανονισμό για το Ταμείο για τι θαλάσσιε δραστηριότητε και την αλληλεία, αλλά η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ικανοποίηση να σα πω, είναι πολύ φιλόδοξη και μπορεί να μα δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με τη μεταρρύθμισή μα. Κλείνοντα, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια σύγκριση με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Χρειάζεται αυτή η σύγκριση. Τη δεκαετία του 90 η αλληλεία των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετώπιζε παρόμοια κατάσταση όπως και εμείς. Όμως το 2007 το Κογκρέσο έθεσε παράνομη, θεώρησε παράνομη την υπερβολική αλληλεία και οι ποσοστώσεις σήμερα τίθενται σύμφωνα με επιστημονική συμβουλή. Σήμερα οι έχουν ουσιαστικά λιγότερη υπεραλληλεία στα αποθέματα από εμά. Μόνο 15%. Εμείς έχουμε 17, έχουν 15. Οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε. Δεν είναι κακοί στο συγκεκριμένο θέμα. Στο συγκεκριμένο θέμα. Ε δεν έχουμε επιλογή παρά να πετύχουμε κι εμείς. Σαν μεγάλη αληφτική δύναμη απλώς δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Θα πρέπει να προσφέρουμε ένα μέλλον για τις θάλασσές μας, για τις βιομηχανίες μας και για τις παράκτιες κοινότητές μας. Ελπίζω ότι με τη βοήθειά σας και με τις γνωμοδοτήσεις σας μπορούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Δαμανάκη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα δώσω αμέσως το λόγο στις πολιτικές ομάδες, στους συντονιστές πρώτα απ' όλα για τρία λεπτά. Και μετά έχω ανοιχτό κατάλογο μιλητών, όποιος θέλει να σημειώνει. Χάκτον, Αρσένης, Βαρέα, Νέβες, Ρέιμερς Λοιπόν, όποιο θέλει να σημειώνει το όνομά του, να σηκώνει και Σάντσα Πρεσέδο, Ρωμέβα, Μιλάνα. Κλείνω τον κατάλογο τώρα όμω. Σας έχουμε, τους συντονιστές τους έχουμε ήδη συμπεριλάβει στον κατάλογο. Δεν τους ανέγνωσα. Τρία λεπτά λοιπόν ο συντονιστής από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τη, και τη Γενική Διεύθυνση για τη δουλειά που έκαναν και μας επιτρέπει σήμερα να έχουμε την παρουσίαση του πακέτου ε, των μεταρρυθμίσεων. Δεν είχαμε ακόμα το χρόνο, εγώ τουλάχιστον είχα το χρόνο να διαβάσω το κείμενο λεπτομερώς, διότι μόνο σήμερα κατέφθασαν μέσω email τα κείμενα, Άρα θα μπούμε στις λεπτομέρειες ε, αργότερα, σε άλλη φάση. Σίγουρα είναι ότι από τις ανακοινώσεις που βλέπω που έκανε η Επίτροπος θεωρώ ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο. Από αυτά που μας είπε μόλις τώρα θεωρώ ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ε, νομίζω ότι η ιδέα της για περιφερειοποίηση μπορεί να λειτουργήσει δίνοντας από ό,τι κατάλαβα μεγαλύτερο χώρο στα κράτη-μέλη ε, αν θέλει να δώσει στα κρατη μέλη και στι περιφέρειε Ευρωπαϊκή Ένωση χώρο και στι κοινότητε φαίνεται σαφές ότι το βέλτιστο είναι εχθρός του καλού. Λοιπόν, ας αρκεστούμε στο καλό, γιατί μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε. Η κοινή πολιτική της Αλίας ε, θεωρήθω σαν εχθρός από πλευράς των αλλιέων μας και όχι σαν κάτι ευχάριστο. Όπως εσείς ανακοινώσατε τα πράγματα, η πορεία αυτή ε, δείχνει ότι μπορεί να λειτουργήσει το, το μέτρο που προτείνεται. Οι ιδιαιτερότητες των θαλασσών ε, τις αναφέρατε εσείς η περιοφυριοποίηση είναι ιδεώδης λύση. Περιμένουμε λοιπόν από αυτή την έποψη ένα καλό αποτέλεσμα. Εγώ ανησυχώ όσον αφορά το θέμα των ποσοστώσεων και των παραχωρήσεων μεταφοράς δυνατότητας αλίας, των εκχωρήσεων που γίνονται αδιάκριτα. Άκουσα, αν κατάλαβα σωστά, ότι δεν θα μπορούν να μεταφέρονται παρά μόνο εντός του εσωτερικού του κάτω μέλους και δεν θα μπορούν να μεταράσουν σε ψαρά Πολύ ασαλία. Γνωρίζουμε όμω ότι ε, υπάρχουν και παγίδε που δεσπίζονται οι νόνοι. Μία τρίτη πρόταση θα ήταν μία περιοριστικός αριθμός εκχωρήσεων που θα μπορούν να μεταφέρονται. Διότι αν αφήσουμε τη δυνατότητα μεταφοράς, πώς να το πω, αυθαίρετη, χωρίς ένα μπλοκάρισμα αριθμητικό, περιορισμό αριθμητικό, μπορούμε να τρέξουμε τον κίνδυνο να υπάρχει ένα μονοπόλιο από πλευράς κάποιων. Ξέρουμε πολύ καλά πώς μπορεί κανείς να ξεγελά τον νόμο. Μπορούν να οργανωθούν εταιρείε που αρχίζουν να αγοράζουν από του ομονωμένους αλληλεί τα δικαιώματα και στο τέλο, δεν θα εφαρμόσουν αυτό που θέλετε. Λοιπόν, ε, εγώ συμφωνώ εν γέννη με τι γραμμέ. Εγώ είμαι πιο σοσιαλιστής από τους σοσιαλιστές θα έλεγα όσον αφορά αυτό το θέμα και πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι μπορούμε να ευνοήσουμε μεγάλες βιομηχανικούς ομίλους και τους μεμονωμένους αλληλείς να τους φέρουμε στη δυσκερή θέση. Αυτό θα το συζητήσουμε όταν ε, θα εκφραστώ καλύτερα όταν θα συζητήσουμε περαιτέρω τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ευχαριστώ. Για τρία λεπτά η κυρία Ρόντους από τους Σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συγχαίρω την Επίτροπο για το έργο που μας παρουσίασε. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο και ξέρω ότι έχουν γίνει και πολλές προσπάθειες και στο παρελθόν. Και από τη νομική υπηρεσία έχουμε ακούσει πόσε δυσκολίε έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Και τώρα για μα ξεκινάει πραγματικά η εργασία στο Κοινοβούλιο από πολλές πλευρές αναμένεται ότι οι ευρωβουλευτές σαν μαριονέτες θα εκπροσωπούν τις εθνικές τους κυβερνήσεις. Αυτό το περιμένουν αυτοί που δεν γνωρίζουν καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι υπεραμεινόμεθα της Ευρώπης και των ιδεών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι αντίβαρο έναντι των εθνικών ε, εγωισμών στο Συμβούλιο. Θέλουμε να παρετηθούμε από τους εθνικούς εγωισμούς και δεν θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε γερμανικούς ή ιρλανδικούς ή ισπανικούς στόχους, θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν είμαστε έτοιμοι να αμφισβητήσουμε και την ίδια τη δική μας θέση όταν βλέπουμε ότι υφίστανται λόγια αμφισβήτησης. Αρκεί να ακούμε τους άλλους και αρκεί να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε συμβιβαστικές λύσεις στα πλαίσια ε, των προπολογισμών που προτίθεται. Νομίζω ότι η πρόταση αποτελεί ένα καλό σημείο θετηρία πάνω στην οποία θα πρέπει να δουλέψουμε εντατικότερα. Και βέβαια πολύ συχνά ο διάβολο βρίσκεται στι λεπτομέρειε, διότι πολλέ προτάσει χρειάζονται μια λεπτομερέστερη ανάλυση. Χαίρομαι γιατί δίνεται μια νέα ε, προσπάθεια, μια νέα όση στην οικολογική διαχείριση και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει ένα σαφή στόχο και δίνει μια νέα όθηση. Αυτό θέτει υποποίηση και τις αρχές των κρατών μελών. Θα πρέπει ε, να ε, ε, θεωρήσουμε θετική αυτή την πίεση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με αυτή τη μεταρρύθμιση να φέρουμε και μια αλλαγή νοοτροπίας και χαίρομαι που αναφέρεται η κατάργηση των απορρίψεων γιατί πραγματικά είναι ένα από τα μέτρα τα οποία πολύ προσεκτικά θα πρέπει να εξετάσουν όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την περιφερειακή προσέγγιση, ξέρω ότι η Επιτροπή αρχικά ε, ήθελε περισσότερα. Ίσως μπορέσουμε να αποκομίσουμε τελικά περισσότερα από την κοινή μας προσπάθεια. θεωρώ ότι η πρόταση τη Επιτροπή αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα και πρέπει να το υποστηρίξουμε. Αναφέρω μόνο τα βασικά σημεία και δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Και τώρα περνάω στις ερωτήσεις προς την Επίτροπο. Υπάρχουν μη διαπραγματεύσιμα ε, ποσοστώσεις ε, ή διαπραγματεύσιμα δικαιώματα και τι ακριβώς σημαίνει. Και τι γίνεται με τις υφιστάμενες ελευτικές δυνατότητες και πώς θα ε, απαλληθούν αυτές. Και άλλη μια ερώτηση σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια. Τι ακριβώς θα συμβεί. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Ευχαριστούμε κύριε Ρόντος. Ε, για τους ελευθέρους ο κύριος Γκάλεχερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω την Επίτροπο και να την ευχαριστήσω που μοιράστηκε μαζί μας ε, τις προτάσεις. Θα ήθελα βέβαια να μην είχαν κυκλοφορήσει πρώτα στα μίντια. Τέλος πάντων, ε, δυστυχώς έτσι συνέβη. Ελπίζω στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. η Κομισιόν λέει ότι είναι πρώτη φορά εδώ που θα και χαίρομαι και με ευγνώμων που υπάρχει στην απόφαση γιατί νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν ε, μείζονε αλλαγέ στι προτάσει αυτέ στου επόμενου 12 μήνε. Θα έπρεπε λοιπόν να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλιο. Σε ό,τι αφορά τι μεταβάσιμε ποσοστώσει, η αρχή ε, με βρίσκει σύμφωνο και ίσω και σε κάποιε χώρε να είναι ε, μια σωστή προσέγγιση. Αλλά σε εμά το 80% είναι κάτω από 15 μέτρα μήκο 80% των σκαφών μα και στην Ιρλανδία δεν θα το δεχθούμε αυτό το μέτρο. Όταν θα έχουμε μεγάλε ευρωπαϊκέ εταιρείε να έρχονται στην Ιρλανδία. σω βραχυπρόθεσμα θεωρηθεί ελκυστικό να πωλήσει, να πωλήσει κανεί ε, ή τέλο πάντων να πάρει ένα δάρ. Δεν ξέρω πώ ε, θα το κάνουμε, αλλά μακροπρόθεσμα θα αποδειχθεί ότι είναι πολύ κακή ιδέα. Ω Κοινοβούλιο και ω Επιτροπή δεν θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ε, ρυθμίζουμε την αγοραπολισία ποσοστώσεων. Και σε ό,τι αφορά τι απορρίψει, πράγματι είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, αλλά και με έναν άλλο τρόπο. Δεν θα πρέπει να είμαστε λαϊκιστές και δημαγωγικοί. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι δεν θα πρέπει τις παρατηρήσει μα να τις ε, επικεντρώνουμε σε κάποιες ε, πολύ συγκεκριμένες ε, εμβληματικές περιοχές αλλά πρέπει να μιλάμε για τους μικρούς αλείς. Δεν θέλουμε να είμαστε αρεστοί και λαϊκιστές αλλά να κάνουμε το σωστό. Πάντοτε κυρία Επίτροπε θαύμαζα τις ε, απόψεις σας σε σχέση με την περιφερειοποίηση. Δεν νομίζω όμως ότι οι απόψεις σας τελικά αντικατοπτρίζονται στην πρόταση που μας παρουσιάσατε. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες νομικές πτυχές, αλλά υπάρχει μια ισχυρή πολιτική βούληση. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας, ώστε να ε, μην υπάρξει αυτή η πολιτική one size fits all, δηλαδή ένα μέγεθος για όλα. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσως ε, αυτό που ισχύει για τη Σκωτία, για την Ιρλανδία, να μην ισχύει για τη Βαλτική, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι η βάση εργασίας για εμάς. Χαίρομαι επίσης που αναγνωρίζονται οι περιφέρειες ε, σας είπα για το μήκος ε, των ε, σκαφών. Εγώ θα προτιμούσα τα 15 μέτρα, αλλά ε, κάποιοι άλλοι μπορεί να πούν κάτι διαφορετικό. Ε, μιλώ για τις παράκτης περιοχές. Πριν καταλήξουμε σε συμπεράσματα, το σκεφτούμε πάντως. Φαίνεται ότι κάποιοι είχαν προετοιμάσει τις προτάσεις τους σε πολύ καιρό. Σας δείχνω κάτι για να δείτε τι εννοώ. Επίσης, έλεγχοι και κυρώσεις, αγαπητή κυρία Επίτροπε, θέλω να ακούσω την άποψή σας ε, επ' αυτών. Αν κάποιος ε, παραβιάσει έναν ε, ελάσσονα κανονισμό, και τελικά του επιβάλλονται κυρώσει αν ήταν εγκληματία. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό. Θα ήθελα να πω και άλλα, αλλά δυστυχώ δεν είχα πάνω από τρία λεπτά. Η πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Λέω για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσίαση που μας έκανε. Κυρία Επίτροπε, πραγματικά περιγράψατε πάρα πολλά και σημαντικά στοιχεία. Και βέβαια τα στηρίζουμε, αυτό είναι προφανές. Στηρίζουμε την απαγόρευση των απορρίψεων, αλλά όταν διαβάσει κανείς το κείμενο, στο βασικό κανονισμό, δυστυχώς δεν μιλάμε για πλήρη απαγόρευση των απορρίψεων ουσιαστικά περιορίζεστε σε κάποια είδη, ε, σε κάποια συγκεκριμένα ψάρια, σε κάποια εμπορικά είδη συγκεκριμένα. Πώς λοιπόν θα εφαρμοστεί η όλη διαδικασία και πώς θα ελέγχεται εάν ε, απορρίπτονται από τον Αλία κάποια είδη και αν κάποια άλλα τα διατηρεί στο σκάφος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Επίσης για το 2015, ναι, πράγματι υπάρχει αυτή η διεθνής υποχρέωση και σίγουρα πρέπει να επιδιώξουμε αυτό το στόχο. Επίσης, η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης ε, πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό υπήρξε πρόβλημα κατά το παρελθόν μας. Ε, δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι στην ανάλυση της Κομισιόν επανειλημμένος από το 2002 και εξή και στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση του 8 και στην πράσινη βίβλο του 2009 Μα δυσαρεστεί το ότι δεν υπάρχει σωστή εράρχηση προτεραιοτήτων μεταξύ των στόχων τη κοινή αλληλευτική πολιτική περιβάλλον, κοινωνική πτυχή, οικονομική στόχη μπαίνουν όλα μαζί στο ίδιο επίπεδο και αυτό υπήρξε η αιτία των συμβιβασμών που είχαμε κατά το παρελθόν. Πώς θα υπερβούμε αυτή την ε, φάση η Κομισιόν ε, λέει διάφορα καλά και επενεί την Αμερικανική νομοθεσία. Τελικά εδώ ε, η παράνομη αλληλεία γίνεται νόμιμη. Δεν υπάρχει επιλογή. Όταν κάποιο πρέπει να επιλέξει μεταξύ βραχυπρόθεσμων οικονομικών ε, κερδών και μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών, κοινωνικών κερδών από την πλευρά της βιωσιμότητας, τι θα προτιμήσει τελικά. Νομίζω ότι πρέπει κάπως να το δούμε γιατί τελικά θα επικρατήσουν τα εμπορικά συμφέροντα. Και να πω και κάποια λόγια στους συναδέλφους μου εδώ από την Επιτροπή. Γνωρίζουμε ότι αυτή η πρόταση θα αποδυναμωθεί από τις δυνάμεις που δρούν εντός του Συμβουλίου. Γιατί το Συμβούλιο ενδιαφέρεται για τα εθνικά συμφέροντα μόνο. Και συμφωνώ με την κυρία Ρόντου. Εμεί εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει το μέλλον όλων των Ευρώπαιων πολιτών, όχι μόνο των αλλιέων σήμερα στις διάφορες χώρες. Μας ενδιαφέρει η ευημερία ε, και η καλή κατάσταση των θαλασσών, των ωκεανών, που είναι πάνω από το ίμιση ε, που καλύπτει πάνω από το ίμιση της επιφάνειας του πλανήτη μας. Και όταν μιλάμε για την βιωσιμότητα των υδάτων, πραγματικά θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε ε, σε σχέση με την έκθεση αυτή και να μην συμπεριφερθούμε ανεύθυνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τρία λεπτά τώρα ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρέπει να γίνει πιο εμπεριστατωμένη μελέτη και πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση. Αλλά Υπάρχουν τρία θέματα που θα ήθελα ήδη από τώρα να τα αναφέρω. Καταρχήν, οι μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις. Αλλάξατε το όνομα, αλλά ουσιαστικά ακριβώς ίδια παραμένει η πραγματικότητα, δηλαδή μεταβιβάσιμο ατομικό δικαίωμα. Επανερχόμαστε δηλαδή με μια ιδέα του 2002, την οποία είχαν απορρίψει τα περισσότερα κράτη-μέλη. Και οι λόγοι που είχαν κάνει τα κράτη-μέλη να απορρίψουν την ιδέα αυτή παραμένουν επίκαιροι κατά τη γνώμη μου. Διότι στην πρόταση της Επιτροπής δεν υπάρχει τίποτα που να μας επιτρέπει να αποφεύγουμε τις αρνητικές συνέπειες ενός τέτοιου συστήματος της μεταβίβασης των ποσοστώσεων δηλαδή. Θα έχουμε μια συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον τομέα. Και αυτό το βλέπουμε στα σημεία που μας ανέφερε η Επίτροπος. Μας είπε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συγκέντρωση. Είπε ότι μπορούμε βέβαια να παρουσιάσουμε διαφορετικά μέτρα για να εμποδίσουμε τη συγκέντρωση. Στο τέταρτο σημείο αναφέρθηκε σε αυτό. Περιορισμένη δυνατότητα μεταφοράς. Παραμένει όμως υποχρεωτικό για τα σκάφη άνω των 12 μέτρων. Και εσείς αναγνωρίζετε λοιπόν, Επιτρόπε, ότι είναι ανεπαρκή τα μέτρα αυτά και θα χρειαστούν νέα μέτρα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη συγκέντρωση στον τομέα. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες τι είδους μέτρα έχετε στο νου σας να λάβετε επιπλέον. Δεν εμποδίζεται η συγκέντρωση ακόμη και με τη λήψη των μέτρων που αναφέρατε. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και εθνικά όρια. Υπάρχει ένα πλαίσιο αγοράς, ε, πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά τρόπον ώστε τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να έχουν ε, ε, σημαντικά ποσοστά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τη συγκέντρωση και πιστεύω ότι και οι άλλες πολιτικές ομάδες που στο παρελθόν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις θα συμφωνήσουν με όσους σήμερα δηλώνουν ότι έχουν αντίρρηση. Η Επιτροπή αναγνωρίζει το πλεονέκτημα του να έχουμε αποκλειστικές ζώνες αλίας με την διατήρηση του ορίου των 12 μιλίων, γιατί η ζώνη αυτή έχει πλεονεκτήματα. Θέλουμε να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση και στις γειτονικές ζώνες πέραν των 12 μιλίων και Η Επιτροπή πολλές φορές έχει δηλώσει ότι χρειάζονται εμπεριστατωμένες επιστημονικές μελέτες. Επί τη βάση των γνωμοδοτήσεων που ήδη έχετε, έχετε λάβει υπόψη την κατανομή των ζωνών στι στις Αζόρες, παραδείγματος, την υφαλοκρηπίδα. Κύριε Στίβενσον, ε, σας πήδηξα <laughs> εντός εισαγωγικών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν ε, ε, σας πρόσεξα. Έχετε τρία λεπτά το λόγο εκ μέρους της ομάδας την ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ και ο Σκεμπάτσεκ, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα αυτά που είχε να μας πει η κυρία Επίτροπος, αλλά βεβαίως πολλές φορές Κυρία Δαμανάκη, σας ακούσαμε να λέτε ότι θέλατε ριζική μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ότι θέλατε περιφερειοποίηση που θα έχει νόημα, αλλά ότι πολεμούσατε ε, μεγάλη μάχη και χρειαζόσασταν βοήθεια. Ε, με λύπη μου λέω ότι εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια. Από αυτά που ακούω και από αυτά που διάβασα μέχρι τώρα, οι γραφειοκράτες φαίνεται ότι νίκησαν τη μάχη. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα μας, μας παραδίδατε μια φάλαινα και σας παραδώσατε τελικά μια σαρδέλα. Το να μας δείτε ότι η περιφερειοποίηση συνεπάγεται να δίνει την υπέροχη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν σε ε, μάτι δικτύων, το μέγεθος του ματιού δικτύου, το έχουν αυτή τη δυνατότητα τώρα. Και θα μπορούν να αποφασίζουν επίσης ε, επί πολιτικών για τις απορρίψεις. Τι, τι γίνεται με το καλάθι των επιλογών που μας υποσχέθηκαν τι γίνεται με το φόρο, με τις ποσοστώσεις, μέρες στη θάλασσα, το σύστημα πιστώσεων για τους αλληλείς, ποσοστώσεις αλλιευμάτων, όλο αυτό το καλάθι των επιλογών. Και εκεί τα κράτη με Έλληνες επιστήμονες εμπλεκομένους στους αλληλείς θα μπορούσαν να διαλέξουν το καλάθι την καλύτερη λύση για τις δικές τους ανάγκες. Εξαφανίστηκε, έλειωσε το καλάθι. Δεν το βλέπω στο κείμενο. Ίσως να κάνω λάθος, ελπίζω να κάνω λάθος αλλά επανειλημμένα. Μας είχατε πει και σήμερα μας το είπατε ότι προσπαθήσατε να πετύχατε λιγότερη μικροδιαχείριση από τις Βρυξέλλες. Όλοι μας εδώ ε, υποστηρίζουμε το να πετύχουμε το μέγιστο επίπεδο, βιώσιμο επίπεδο ε, αλίας μέχρι απόδοσης μάλλον του 2015. Αυτό προσπαθούμε δεκαετίες, αλλά μας έχει παιδέψει η μικροδιαχείριση από τις Βρυξέλλες. Αυτό μας εμπόδισε. Ο στρατός των γραφειοκρατών. Έχει εισαχθεί αυτή πληθώρα ε, κανόνων, κανονισμών ε, που δημιούργησαν ένα χάλι, το είπατε επανειλημμένα, καταστροφική κατάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, αλλά φαίνεται ότι εδώ τελικά παγιώνεται, προστατεύεται, ε, θα συνεχίσει. Εγώ νομίζω πραγματικά ότι αυτή η πολιτική που έχετε παραγάγει είναι μέτρια, μετριοπαθής και το λέω ευγενικά αυτό. Δεν θα χρησιμοποιήσω κάποια ισχυρότερη διατύπωση που μ' ακούνε να λέω στο γραφείο μου, πιο ισχυρές εκφράσεις. Πάντα είστε πολύ ευγενείς. Πάντα είστε ευγενείς εδώ, κύριε Στίβος. Λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε στους συντονιστές ή να δώσω σε όλους πρώτα το λόγο και να... Εσείς επιλέγετε, εσείς είστε οι προσκεκλημένοι μας, ε, δεν θα αποφασίσω εγώ, λέει πρόεδρος. Ωραία, το κανονίσαμε. Λοιπόν, 15 έχω σημειώσει και κλείνω τον κατάλογο αν θέλετε να απαντήσει και να έχει χρόνο η Επίτροπος σε όλους, μην υπερβείτε το ένα ε, λεπτό, ε, ώστε να μπορέσει να έχει χρόνο η Επίτροπος. Τους άλλους και οι συντονιστές μίλησαν εξ ονόματό σας. 15. Επί ένα λεπτό, 15 λεπτά. Κάπου τόσο τα υπολογίζω, για να έχει χρόνο και επίτροπος. Λοιπόν, κυρία Τότ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε να μας δείτε σήμερα. Εγώ θα αναφέρω τρία βασικά θέματα, αποκέντρωση όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και τις απορρίψεις. Για την αποκέντρωση συμφωνώ με τον Στρούαν Στίβενσον. Νομίζω ότι εν γέννη είμαστε απογοητευμένοι. Θέλουμε να δούμε πραγματική πρόοδο και δεν θέλουμε να δούμε αποκέντρωση που να έχει αποδυναμωθεί τελικά στις ε, διαπραγματεύσει πολιτικέ που λαμβάνουν χώρα εδώ. Όσον αφορά τι απορρίψει, όλοι συμφωνούμε ότι οι απορρίψει είναι κάτι κακό, δεν είναι καλό για τα αποθέματα, για τη βιομηχανία και δεν το θέλουν οι καταναλωτέ. Πρέπει να πω ότι αυτό που δεν θέλουμε είναι να δούμε την πρόοδο που ήδη πετύχαμε εντό του τομέα να πεταχθεί να πάει χαμένη λόγω τη πιέσεω των μέσων ενημέρωση. Θα πρέπει να θυμόσαστε ότι η πρόοδο εμποδίζεται από το εξή γεγονό ότι τα παρόντα οικονομικά μέτρα σημαίνουν ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε ταχύτητα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε να αλλάξουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιείται στην αλληλεία που θα βοηθούσε στη μεικτή αλία που λαμβάνει η χώρα σε θάλασσε όπω είναι η Ιρλανδική θάλασσα. Πολύ γρήγορα να πω κάποια πράγματα. Πρέπει να δούμε στοιχεία, περισσότερα στοιχεία και να τονίζονται περισσότερο τα στοιχεία και τα λεφτικά αποθέματα. Ε, πολλά από τα αποθέματα θεωρείται ότι δεν δίνουν επαρκή στοιχεία και χρειαζόμαστε τους πόρους πόρου για να συλλέγουμε στοιχεία. Σας ευχαριστώ κύριε Αντότσο. Κύριο Χάγκλουτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσία της, για την παρουσία της εδώ. Θα επικεντρωθώ σε ένα θέμα, τη μικρή κλίμακα σπαρακτεαλία. Όταν εκπονήσαμε την έκθεσή μας ε, για την πράσινη βίβλα εξαιρετική έκθεση συναδέλφου Πάτρον Νέβες, είχαμε τονίσει την ανάγκη υπαρξής μιας ε, ειδική προσέγγισης για τη μικρή κλίμακα παρακτιαλία. Βλέπουμε τώρα ότι η περιφερειοποίηση όπως τη λένε οι φίλοι από τη Βρετανία, ε, προκαλεί απογοήτευση για πολλούς. Ξέρω ότι το, καθήκον, μάλλον το έργο της Επιτροπής δεν ήταν εύκολο αλλά ε, παρότι δεν ε, είχα χρόνο να μελετήσω το άρθρο, το έλαβα πριν από κάποιες ε, ώρες, βλέπω ότι κάπου ανεπαρκής είναι η αναφορά στην μικρή κλίμακα σπακαλία. Κάπου λείπει, είναι ο κρίκος αλήθως που λείπει. Αν θα θέλετε να σχολιάσετε παρακαλώ. Μπράβο σας κύριε Χάγκλουτ, τηρήσατε το χρόνο. Ο κύριο ε, Καντέκ, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ένα λεπτό όμως τι να πει κανείς, δεν θα είναι απλό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Κάποια από τα μέτρα τα οποία μας παρουσιάσατε φαίνονται ενδιαφέροντα, ωστόσο εγώ δυσκολεύομαι να ε, συμμεριστώ την αισιοδοξία σας για κάποια από τα στοιχεία της μεταρρύθμισης που μας προτείνετε και συγκεκριμένα όπως ξέρετε δεν είμαι υπέρ αυτών των μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων ακόμη και εντός χωρών και ακόμη και με ασφαλιστικές δικλείδες γιατί νομίζω ότι ε, ουσιαστικά έχουμε συγκέντρωση των δικαιωμάτων κάτι που θα είχε δραματικές επιπτώσεις για τη μικρή κλίμακα παράκτη στην Ευρώπη. Ούτε μου αρέσει η ιδέα ε, των μηδενικών απορρίψεων. Καλό θα ήταν να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και να υπάρχει μεγαλύτερη επιλεξιμότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιφερειοποίηση, ελάχιστα κάνει την εμφάνισή της στην πρότασή σας και ε, αυτή την, ε, τους στόχους ε, για την ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015 ε, δεν μου φαίνεται και τόσο πολύ ε, αισιόδοξη ως πρόβλεψη. Πάντως, σε ό,τι αφορά τη σχετική σταθερότητα, εμένα είμαι πολύ κατηγορηματικός. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κούν. Συγγνώμη, απλά για να μην πεθάνουν οι διερμηνείς, πρέπει να τη βγάλουν τη μέρα. Ε, εντάξει, είναι λίγο το ένα λεπτό, αλλά τουλάχιστον ε, να έχουμε ένα μέτρο στην ταχύτητα. Ευχαριστώ κύριο Σκούρ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε με την Ντάουσα θέλουμε να πούμε καλά ή στοιχεία κριτική προ την Επίτροπο. Δεν μα μένει χρόνο να πούμε τα τη ουσία. Όσον αφορά την σχετική σταθερότητα, συμφωνώ και εγώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στον προγραμματισμό. Και τα σχέδια διαχείριση που αναφέρατε, Επίτροπε, για μα είναι εξίσου σημαντικά. Χρειαζόμαστε εκεί ορθολογική διαχείριση, αλλά όχι με τη λογική ότι 25% άρα κόβουμε. Θα πρέπει να γίνει μια σαφή συζήτηση. 15% συν ε, είναι αρκετά τολμηρή πρόταση. Και μπορούμε να πούμε ότι παραμένουμε στα μέγιστα ε, ε, στα τάκ που επί χρόνια τα έχουμε δοκιμάσει ε, και μπορούμε να μειώσουμε την αλληλευτική προσπάθεια και τον αριθμό των ημερών. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι μικρέ επιχειρήσει, οι οποίε παραδίδουν άμεσα φρέσκα ψάρια στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία. Αυτοί πρέπει περισσότερε μέρε να παραμένουν στη θάλασσα. Δεν μπορούν να μείνουν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό κάθε αλληλευτική περίοδο. Όσον αφορά τι απορρίψει, πρέπει να δούμε ποια είναι τα είδη τα οποία απορρίπτονται για να μην χάνονται τα αποθέματα τα οποία πραγματικά χρειαζόμαστε. Και αν μειώνεται το στόλο, πάλι θα πρέπει να γίνει με ειδικευμένο τρόπο ανά κράτο μέλο, Αλλά πρέπει να δούμε πόσα είναι τα τάπια τη Γερμανία και πόσο είναι ο, στόλο. στόλος, που είναι πολύ διαφορετικά τα ποσοστά. Ε, ολοκληρώσατε ή όχι. Γιατί κάποιος ε, σας διέκοψε, ολοκληρώστε ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Wir leben nicht allein δεν είμαστε μόνοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και οι τρίτες χώρες με τις οποίες πρέπει να διαπραγματευτούμε. Γι' αυτό μας απασχολεί ακόμη περισσότερο στις χώρες της Μεσογείου που έχουν επαφές με τις νότιες χώρες ή και στο Βορρά με τη σχέση με την Νορβηγία. Δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε άγιους αυτούς στο Βορρά. Παντού ε, υπάρχουν σχετικά ζητήματα. Μήπως έχω τρία λεπτά και μπορώ να συνεχίσω. Φινίτο λέει πρόεδρος. Ο κύριος Χιούτον. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να κάνουμε πληρέστερη ανάλυση. Λίγα σχόλια μόνο προ το παρόν. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετέ αντιφάσει στο σημερινό έγγραφο στην ανακοίνωση μέχρι τη σελίδα 2, παράγραφο 2, έφτασα όπου λέει ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική έχει τεράστιο δυναμικό για να βοηθήσει για την βιώσιμη αλληλεία. 30 χρόνια εμπειρία έχουμε στην Σκοτία και ακόμη δεν τα έχουμε καταφέρει να ε, επιτελέσουμε αυτό το στόχο και με όσα βλέπω σε αυτό το έγγραφο δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να εκπληρωθεί ο στόχο αυτό στο μέλλον. Η αλληλευτική πολιτική έχει αποτύχει και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μα έχει βοηθήσει να ξεπεράσουμε τη διένεξη για το σκουμπρί που μα δημιουργεί τεράστια προβλήματα προ το παρόν. Είπατε επίση ότι είστε υπέρ τη περιφερειοποίηση, αλλά τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα θα είναι υποχρεωτικά και άλλε αντιφάσει λοιπόν. Είπατε ότι είστε υπέρ της περιφερειοποίησης, αλλά για τις απορρίψεις θα εφαρμόσετε κάποια απαγόρευση ή κατάργηση, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το ονομάσετε. Και αυτό είναι άλλο ένα από τα προβλήματα της μικτής αλίευσης. Στο έγγραφο υπάρχει επίσης ε, στο σημείο 4 η δήλωση προαιρετικά στοιχεία επιβεβαιώνεται η αρχή της ίσης πρόσβασης στα ύδατα και στους πόρους. Εγώ δεν βλέπω πώς θα μπορούσε αυτό το σημείο να δώσει τη δυνατότητα στην περιφερειοποίηση και να μας δώσει την ελπίδα ότι ότι θα μπορούν πραγματικά οι αλληλείς και ιδίω ε, ε, ε, χώρες που βασίζονται στην αλληλεία όπως η Σκοτία θα υποφεληθούν από βιώσιμη αλληλεία και από διατήρηση των ειδών. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αν πρέπει να σας διακόπτω όλους θα βγάλω κάποιους από τη λίστα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο κύριος Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επίτροπο για τα αυτά που μας ανέφερε και όσον αφορά ε, τις, που μετάφρασε διάφορες ιδέες σε δράσεις. Αυτό είναι το θέμα. Ε, να αναφέρω κάποια θέματα που το μη συμφορώ. Το μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Εκεί δεν υπάρχει αντικειμενικός στόχος, λόγος να μας οδηγήσει να υπολοιπόμεθα των υποχρεώσεων του Johannesburg. Λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα στο Johannesburg. Πρέπει να τηρήσουμε και έχουν ληφθεί και αποφάσεις εν ώψη του 2020. Τώρα για τα μεταφερόμενα δικαιώματα ε, δεν συμφωνώ. Αν υιοθετηθεί το μέτρο, η διάταξη θα πρέπει να ισχύει σε κάθε κράτος μέλος, όπως προτείνει η Επίτροπος. Αλλά ε, θα πρέπει να αποφύγουμε συγκέντρωση και συγκέντρωση σε ένα κράτο μέλος. Θα είναι κάτι κακό. Χρειάζεται να είναι θελοντικό το μέτρο. Αυτό θα ήταν ο συμβιβασμός. Λείπουν αναφορές στην υποστήριξη του εξυγχρονισμού. Χρειάζεται υποστήριξη ο εξυγχρονισμό των στόλων, χωρί να σημαίνει αύξηση αλληλευτικού δυναμικού. Χωρί την υποστήριξη θα συμβεί. Είσαστε Ελληνίδα, γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η οικονομική κατάσταση που κρατεί σε πολλά κράτη-μέλη. χωρί κοινοτική βοήθεια δεν μπορούμε να εξυγχρονίσουμε του στόλου μα. Θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή σύμφωνα με την οποία δεν θα αυξήσουμε το δυναμικό τη αλίας. Θα πρέπει όμω να είμαστε ανοιχτοί στη βοήθεια σε εξαιρετικέ περιστάσει. Τόσο αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες, συμφωνώ με τη συγκεκριμένη αρχή ότι θα πρέπει να συνάπτουμε συμφωνίες όταν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ίσως να υπάρχουν καταστάσεις όμως όπου δεν υπάρχουν ε, οι επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες και και θα ξερούμε την δραστηριότητα των στρόλων γιατί λείπει ε, αυτή Επίτροπε, ε, μας περιγράψατε την δραματική κατάσταση των αλληλευμάτων σήμερα, αλλά και ποια θα είναι η κατάσταση το 2022 αν δεν λάβουμε μέτρα. Απαιτείται μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η πρότασή σας, που είναι και ισορροπημένη και εφαρμόσιμη. Αυτό που μου λείπει από την πρότασή σας είναι ότι θα ήθελα μια πιο ξεκάθαρη ε, εστίαση στην οικοσυστημική προσέγγιση. Θα ήθελα μια πιο ξεκάθαρη εστίαση ε, στη σημασία ε, των προτεραιοτήτων που αναφέρθηκαν και από άλλους συναδέλφους, ότι προφανώς πρέπει να έχουμε ψάρια για να μπορούμε να ψαρεύουμε. Επίσης, θα ήθελα να δούμε το θέμα των περιοχών προστασίας εκθαποθεμάτων Περιοχές δηλαδή που δεν ψαρεύουμε προκειμένου να αυξάνεται και να προστατεύουν τα αποθέματα, αλλά και να αυξάνεται η αλία γύρω από αυτές ε, όσον αφορά την, ε, τα discards, θα πρέπει να δούμε το θέμα των, ε, της επιλεκτικότητας των αληφτικών εργαλείων. Είναι κάτι που δεν είδα αρκετά στην πρότασή σας, θα θέλω να το ενισχύσουμε. Και τέλος, για να μην παίρνω το χρόνο των συναδέλφων, ε, θα πρέπει πάντοτε οι αποφάση μας να στηρίζονται στα επιστημονικά δεδομένα και αυτό είναι μια αρχή που σεβόμαστε αυτή την Επιτροπή και θα στηρίξουμε στη μεταρρύθμιση της κοινής αληθικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ κύριε Αντρές Μπαρέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα. Επί της αρχής μας τα παρουσιάσατε τα πράγματα, ε, κάπως ομά, δεν ε, λειτουργήσαν τα πράγματα και στη διαχείριση δεν τα καταφέραμε. Ε, μιλήσατε για αύξηση της περιφερειοποίησης. Εγώ θέλω να τονίσω την αρχή αυτής της περιφερειοποίησης και της διαχείρισης. Δεν μιλάμε για πολιτική αποκέντρωση. Μια Ισπανίδα μιλάει σε μια Ελληνίδα εδώ. Σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για κάθε θέμα, οικονομικό, κοινωνικό και για θέματα βιωσιμότητας. Είναι θεμελιώδες στοιχείο και να μην κάνουμε λάθος, να μην αφήσουμε άλλοι φορείς να λύσουν τα προβλήματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε συνολικά σε επίπεδο 27 χωρών μελών. Σε ό,τι αφορά τώρα τις απορρίψεις, θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό υπό τα κριτήρια του Johannesburg και να μιλήσουμε για την οικοσυστημική ε, εστίαση. Τώρα σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις με τις εκχωρήσιμε, δεν ξέρω αυτό πώς θα το δείτε μέσα στην ενή αγορά γιατί υπάρχει αντίφαση εδώ δεν ε, γίνεται λόγος για την παράκτεια αλληλεία, τη σχέση με τρίτες χώρες και την παρουσία μας ε, ε, μέσω των συμφωνιών που έχουμε σε τρίτες χώρες όπως η Κίνα για παράδειγμα που έχουν αρπακτικές διαθέσεις και δράσεις. Δεν ακούμε αρκετά, δεν έχουμε στην εκθέση πώς και, και πώς, πότε θα ήθελα να μας πείτε. Κυρία Πατράχη τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή αλληλευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτάσεις τις οποίες διέταξαν η συντομία έχουν κάποιες γενικές αρχές αλλά δεν μπαίνουν σε επαρκείς λεπτομέρειες. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα στοιχεία για να μπορέσουμε ε, να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Καταρχήν για την περιφερειοποίηση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα συνδεδεμένες προτάσεις, γιατί εδώ υπάρχει η μεγάλη ακαμψία στις προτάσεις. Με τι μέτρα και σταθμά κρίνεται την υδατοκαλλιέργεια, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει αντίστοιχο περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο. Όσον αφορά τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, ε, θα έχουμε κατά νου την ε, βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ληφθούν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συμφωνίες με την Κίνα. Τέλος, για τον προϋπολογισμό, για να έχουμε μια ισχυρή αλληλευτική πολιτική, χρειαζόμαστε υψηλότερου πόρου. Ενώ είπατε ότι είναι παρόμοιο ο προπολογισμό ε, με την προηγούμενη χρονιά που δεν είναι επαρκέ. Κυρία Ράιμερ, ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Θα περιοριστώ σε πολύ λίγα στοιχεία και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ε, ε, θα πρέπει στο μέλλον όλες οι, όλα τα αλλιεύματα τα οποία προείζουν για απορρίψει να εκφορτώνονται. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα αλλιευτικά αποθέματα. Έχουμε ενδεχομένω κάποιο μικρό απόθεμα για κάποιο είδο, το οποίο ω παρεπίπτον αλλίευμα ε, εξαντλείται, εξαντλείται η ποσόστοση. Οπότε τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, πώς θα ε, επιληθεί το πρόβλημα όταν τα αλλιεύματα δηλαδή, ε, όταν οφείλεται στα αλλιεύματα ο περιορισμός της συνολικής εκφόρτωσης. Ξέρω ότι είναι πολύ πλοκή ερώτησή μου. Κύριε Μπλιμπάου. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε για 75% υπεραλίευση σε ορισμένες περιοχές και ακούσαμε και για τη δεκαετία του 90 και για την μη αποδοτικότητα του κλάδου. Χρειαζόμαστε όμως αριθμητικά στοιχεία για την αλληλευτική δυνατότητα που πραγματικά έχουμε σήμερα πόσα ε, σκάφη έχει ο στόλος, πώς είναι η αλληλευτική ικανότητα. Για να σα πω για το Μερλό και για το Γάβρο, τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν την ίδια τιμή περίπου. Επίση, ό,τι αφορά τη βιομηχανία και τι απώλειε, ασφάλεια των τροφίμων, ε, πλούτο. Τι θα κάνουμε με τη συγκεκριμένη πρόταση, με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, όταν έχουμε καταγγελίε μόνιμε από τον αλληλευτικό κλάδο για προϊόντα τα οποία έρχονται από τι ε, τρίτε χώρε. Και μαζί με αυτό θέλω να μου πείτε αν με αυτή τη μεταρρύθμιση θα αλλάξει ο ρόλο που θα έχει ο λευτικό ε, κλάσο, είτε αφορά χάρη την σύναψη, την υπογραφή εμπορικών συμφωνών. Τρίτο πυλώνα. Μιλάτε για συνέπεια και ε, συνοχή και στον τομέα αυτό. Με τι απορρίψει. Τι λύσει θα έχουμε σε σχέση, παραδείγματο χάρη, με τη μεικτή αλία. Μπορεί να συμφωνούμε με το ένα ή με το άλλο, αλλά Ποιε είναι οι συγκεκριμένε λύσει που προτείνεται για τη μεικτή αλία. Επίση, ε, διακυβέρνηση, περιφερειοποίηση, ναι, μεγαλύτερε ευθύνε και αρμοδιότητε για τον κλάδο. Αλλά όταν έχουμε και αυτά τα πολιετή σχέδια, αυτά τα μακροπρόθεσμα προγράμματα. Τελικά ε, αυτή η δυνατότητα διαχείρισης αυτών των θεμάτων μέχρι που μπορεί να φτάσει, τι θα γίνει με το Συμβούλιο και σε σχέση ε, με τις σχέσεις ε, με τρίτες χώρες και τις συμφωνίες έχουμε σαφή απειλή Κίνα και Ταϊβάν και για την Αλία γενικότερα και για τις συμφωνίες νέας γενιάς που είπατε σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα θα είμαστε συνεπεί και σε σχέση και με άλλου τομεί, Παραδείγματο χάρη αυτοκινητοβιομηχανία, κλωστεφαντουργία ή αυτά για τα, θεμελιώδη, για που θα ισχύσουν μόνο για τι αλληλευτικές συμφωνίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Εγώ εύχομαι στην εμβάθυνση που θα κάνουμε στο έγγραφο να βρούμε τη λέξη απλούστευση. Εύχομαι να βρούμε μια ισορροπία όσον αφορά την οικονομική συνέπεια, τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει αυτή η επιλογή. Διότι δεν θέλω να αντιμετωπίσω το ότι η βιωσιμότητα αντιστοιχεί ακριβώς και απλούς, απλώς μόνο σε μία φάση κυρώσεων ενός μόνο από τους ε, φορείς που ε, συνδράμει στη μείωση της βιοποικιλότητας, στους αλείς και μόνο δηλαδή να επιβάλλεται διότι αν ακολουθήσουμε μόνο αυτή την προσέγγιση και αν αναφέρεται αυτούς τους όρους ε, δεν είναι σωστό, είναι πιο περίπλοκο. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία κάνενο θέματος, θέλω να πω μόνο αυτό. Αν αυτή η πολιτική λειτουργεί σημαίνει απλώς ότι θα υπάρχει λιγότερο ψάρι που θα αλλιεύεται, θα υπάρχει μια οικονομία που θα έχει λιγότερου πόρου, Θα πρέπει να συνοδεύεται αυτό από την έξοδο από αυτό το τομέα εργαζομένων και επιχειρήσεων μέσω της υποστήριξης για αυτή την έξοδο. Δεν θα ήθελα αυτός να είναι ο μόνος τομέας στην Ευρώπη στον οποίο όταν βγαίνει κανείς ε, από τη Χαλιβουργία συνοδεύεται όταν φεύγει και αυτός που φεύγει από την Αλία δεν συνοδεύεται ο Αλίας για να φύγει από τον τομέα. Σενιόρ Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα στα σχόλια που ακούστηκαν. Όσον αφορά την μεταφορά των ποσοστών δικαιωμάτων είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Η συγκέντρωση και η κερδοσκοπία ε, είναι ένας κίνδυνος από αυτή την πρόταση. Πρέπει να εξεταστούν. Από την άλλη πλευρά στην πρόταση δεν βλέπω την το να ζητείτε από τους αλληλείς να δρουν με συγκεκριμένο τρόπο για τη βιωσιμότητα. Πώ ψαρεύουν, ποιο έχει το δικαίωμα να ψαρεύει. Δεν είναι μόνο θέμα τη εμπορία δικαιωμάτων, είναι θέμα ποιο πρέπει να έχει το δικαίωμα να λιεύει και πώ. Ε, και αυτό είναι που θα πρέπει να ε, οδηγεί στην απόφαση το ποιο. Αυτή που είναι πιο υπεύθυνοι όσον αφορά την κατάσταση τη ενέργεια και όσον αφορά τη λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον, αυτοί θα πρέπει να είναι προνομιούχοι εν συγκρίση με τους άλλους, τη μεγάλη βιομηχανία δηλαδή, που πολύ συχνά ψαρεύει με πιο επιζήμιο τρόπο από ό,τι άλλοι. Αναφέρατε μετά και τονίσατε το θέμα των ιδετοκαλλιεργιών Ε, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο θετική. Στη Γαλλικία ε, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο Τουρινιάν, όπου κάποιες εγκαταστάσεις ιδετοκαλλιεργιών είναι στην, εντός του δικτύου Natura ε, αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλος ιδιαίτερος. Και τέλος μια ερώτηση. Τι έγινε με τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, την, την είδαμε σε κάποιες τις προηγούμενες προτάσεις, αλλά εδώ μας λείπει. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο έχει λησμονηθεί ή απλώς εξαλειφθεί κατά κάποιο τρόπο. Αλλά είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση όταν δεν αναφέρουμε τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την διάσταση αυτή. Ε, Ευχαριστώ Σάντσεφ Πρισέδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εγώ Συμφωνώ απόλυτα ότι βασικά η αρχή που θα διέπει τη μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι η βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά τα ατομικά μεταβιβάσιμα δικαιώματα. Ε, πώς θα προσαρμόσουμε τις αλληλευτικές δυνατότητες στους πόρους ε, αν δεν έχουμε την απαιτούμενη ευελιξία και αν συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή την τόσο άκαμπτη διαχείριση ε, των πόρων. Θέλω να σας θέσω τα εξή ερωτήματα. Πρώτον, θα υπάρξει διαφοροποιημένη μεταχείριση της μικρής κλίμακας παράκτειας αλίας. Αυτό είναι σημαντικό ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Θα γίνει μια πλήρης μεταρρύθμιση που θα περιλαμβάνει και την ε, υδατοκαλλιέργεια, ε, άρα συμφιλιώντα υδατοκαλλιέργεια και περιβάλλον. Και τρίτον, ε, συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς και συνεκτικοί. Άρα, οι εξωτερικέ συμφωνίε θα πρέπει να βασίζονται στην ίδια αλληλευτική πολιτική με αυτή που εφαρμόζουμε εμεί εδώ. Αλλά το ίδιο θα πρέπει να ισχύει στι εισαγωγέ. Δηλαδή, θα, ρωτώ, θα είναι τα ίδια κριτήρια και για τι εισαγωγέ. Ευχαριστώ, κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέντε σύντομε παρατηρήσει για τι μεταβιβάσιμε ε, ποσοστό αλληλεία. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Είναι νέο όνομα για αυτό που ονομάζουμε ποσοστώσει με εντελώ διαφορετικέ διατάξει. Δεύτερον, το 20% των αλληλευτικών αποθυμάτων βρίσκονται ε, κοντά στην ε, περιοχή, που βρίσκονται κοντά στην περιοχή τη Ιρλανδία, υπεραλλιεύονται και όχι από Ιρλανδού αλληλεί και θα ήθελα επίση να πω ότι έχω μεγάλο πρόβλημα με την περιφερειοποίηση, γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε τα ίδια μέτρα ε, με τον ίδιο τρόπο παντού. Δεν μπορούμε να έχουμε μια αλληλευτική πολιτική την οποία θα εφαρμόζουμε διαφορετικά ε, ε, αλληλευτικά μέσα. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνταχθούν εκ νέου πολλά από αυτά τα μέτρα, γιατί τα περισσότερα δεν τα θεωρώ αποδεκτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο και δεν έχει λάβει το λόγο. Όχι. Άρα κανείς δεν είναι παραπονεμένος. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για το ενδιαφέρον τους και για τις απόψεις που εξέφρασαν. Θα ήθελα να εξηγήσω το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα δεν επανέρχομαι πάλι ε, για να ξανασχεδιάσουμε την πολιτική από την αρχή όπω πρότεινε κάποιο ομιλητή. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε ε, στο πλαίσιο τη συναπόφασης να συζητήσουμε με βάση τι τροπολογίε σα για να συζητήσουμε και να βρούμε την καλύτερη λύση για όλα τα προβλήματα. Ε, ίσως παρατηρήσατε κάποια προβλήματα, μερικά από αυτά μπορεί να υπάρχουν, άλλα μπορεί να μην υπάρχουν αλλά είναι προφανές ότι επιμένετε σε πολλές από τις απόψεις σας και πολλές ε, από τις απόψεις σας είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Υπάρχουν βουλευτές που μίλησαν υπέρ μιας πιο ριζικής μεταρρύθμισης για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Άλλοι θεωρούν ότι προχωρούμε υπερβολικά γρήγορα. Κάπου πρέπει να τηρήσουμε μια ισορροπία και πρέπει να συνεργαστούμε με όλα τα γραφεία ε, των επιτρόπων, με όλους τους επιτρόπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, χαίρομαι διότι υπήρχε ε, ομοφωνία σήμερα και είναι πολύ θετικό το να έχουμε θετική υποστήριξη σε ομοφωνία από την Επιτροπή. Εγώ είμαι εδώ για να συνεργαστώ μαζί σας και είμαι ιδιαίτερα πρόθυμη να δεχθώ τις προτάσεις σας στις οποίες θα καταλήξουμε. Χρειάζεται περισσότερη συζήτηση και καταλαβαίνω ότι θέλετε να δείτε και τις λεπτομέρειες. Και σίγουρα θα πρέπει να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες και νομίζω ότι θα βρούμε τον τρόπο ε, για να ξανά έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί. και οι υπηρεσίε μου θα μπορέσουν να σα δώσουν και λεπτομερεί απαντήσει σε όλε σα. Να σα δώσουμε λεπτομερεί απαντήσει όσον αφορά το κείμενο αφού το κείμενο σήμερα δημοσιεύθηκε δεν έχετε ακόμη ενημερωθεί πλήρω. Θα ήθελα να σχολιάσω ε, κάποιες από τις παρεμβάσει σας, όπου έχω να σα δώσω κάποιες διευκρινήσει, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχετε και τις δικές σας απόψεις σε πολλά θέματα. Ε, καταρχήν για την περιφερειοποίηση. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, παραμένοντας συμβατοί με τις συνθήκες μου είπατε πολλοί από εσά ότι έχετε απογοητευτεί και θα ήθελα να εξηγήσω πλήρως τη θέση μας. Εδώ μπορούμε να δεχθούμε τροπολογίες που θα εμβαθύνουν αυτή τη διαδικασία, που θα ζητήσουν κάτι περισσότερο φιλόδοξο για την περιφερειοποίηση υπό έναν όρο, ότι η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου θα μου δώσει μια γνωμοδότηση ότι αυτό είναι συμβατό με τη συνθήκη. Εάν μου το δώσετε αυτό, μπορούμε να συνεργαστούμε και να το συμπεριλάβουμε. Αλλά φοβούμαι ότι ορισμένε από τι προτάσει σα αντιβαίνουν προ τι συνθήκε άμεσα. Παραδείγματο χάρη, αν λέτε ότι οι ποσοστώσει πρέπει να μεταφέρονται ε, σε περιφερειακούς οργανισμούς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε λόγω της συνθήκης. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μιλάτε για τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης. Ας αφήσουμε τη συνθήκη κατά μέρο και να σας ρωτήσω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Αλληλείας του Κοινοβουλίου, κυρία Πρόεδρε, είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει την αρμόδιότητά της ε, να, αποφασ... να παραιτηθεί ε, από τους ε, από την αρμοδιότητά τους για, του, για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα και να το δώσει σε περιφερειακούς οργανισμούς. Νομίζω ότι δεν είστε ούτε εσεί ε, υπέρ αυτή τη άποψη και γι' αυτό σα παρακαλώ να είστε όλοι λογικοί και να καταλάβετε ότι εδώ έχουμε κάποιε δεσμεύσει που πρέπει να τηρήσουμε. Πρέπει να σεβόμεθα τη συνθήκη και δεν μπορούμε να υπερβούμε τη συνθήκη. Καταλαβαίνω ότι ενδέχεται να έχουμε κάνει λάθη και πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση, να δούμε αν υπάρχει κάποιο περιθώριο, να δώσουμε μεγαλύτερη αρμοδιότητα στα περιφερειακά συμβούλια. Ε, και ειλικρινά ε, το εννοώ αυτό που λέω, ότι θα είμαι εδώ και θα συνεργαστώ μαζί σας εάν μου δώσετε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου ότι αυτό το οποίο μου ζητάτε είναι συμβατό με τη συνθήκη. Είμαι υπέρ της περιφερειοποίησης όπως και εσείς. Σας διαβεβαιώ, γιατί αυτό το παζάρι το έχω ζήσει στο Συμβούλιο και είναι εφιάλτης, δεν θέλω να το ξανακάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Κυρία Ντότς, αναφέρατε τα Ιρλανδικά σκάφη ε, και αλληλευτικό εξοπλισμό. Μπορούν τα περιφερειακά συμβούλια να γνωμοδοτήσουν και να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε. Αναφέρεται τα μεγέθη των ματιών των δικτυών. Αυτό δεν είναι απλώς λεπτομέρεια, αν το μέγεθος των ματιών των δικτυών και όλα τα τεχνικά μέτρα αποτελούν ε, απλή λεπτομέρεια και το να ε, κλείνουμε τον τομέα για δύο μήνες κλπ. Δεν είναι λεπτομέρειες. Διαφορετικά γιατί μου στέλνετε αποστολές. Δεν είναι καθόλου λεπτομέρειες. Είναι σημαντικά ζητήματα. Ίσως δεν είναι επαρκή αυτά που προτείνουμε και πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, αρκεί να βρούμε προτάσεις συμβατές με τη συνθήκη. Και επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι που το εννοώ και ξέρετε ότι είμαι απόλυτα ειλικρινής. Νομίζω ότι με γνωρίζετε πλέον. Τουλάχιστον ειλικρινής είμαι ό,τι ελαττώματα άλλα και αν μου προσάπτετε. Τώρα, για, τις, για τα δικαιώματα. Και αυτό είναι αντιφατικό θέμα και θα χρειαστούν πολλές συζητήσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Να σας εξηγήσω όμως αυτά τα οποία τώρα περιλαμβάνονται στο κείμενο και μετά αν θέλετε υποβάλλετε τροπολογίες για να αλλάξουμε αυτά που υπάρχουν στο κείμενο. Μιλάμε για μεταβιβάσιμα δικαιώματα. Ε, τι θα γίνει με την παράκτια αλία μικρής κλίμακας. Μπορούν τα κράτη-μέλη να δώσουν απαλλαγές. Ο κύριος Σάντος που αναφέρθηκε ε, στην Πορτογαλία ε, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που συζητάμε για τα δικαιώματα αφορά το 16% των σκαφών σας μόνο. Η κατάσταση στην Πορτογαλία έχει ως εξής. Το 16% είναι πάνω από 12 μέτρα, αλλά παίρνουν το 90% ε, της συνολικής, ε, του συνολικού δυναμικού. Ε, μιλάμε λοιπόν μόνο για τα μεγάλα σκάφη όταν μιλάμε για, τις, για τα δικαιώματα. Και τα κράτη-μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν περισσότερες ρήτρες διασφάλισης και μου μιλήσατε για τον κίνδυνο της συγκέντρωσης, τον οποίο ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε. Πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να φροντίσουν αν ένα παραγαδιάρικο έχει κάποιο δικαίωμα να μπορεί να το πουλήσει μόνο σε παραγαδιάρικο και όχι σε μικρότερο σκάφος. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι μπορείτε να πουλήσετε δικαιώματα μέχρι κάποιο επίπεδο. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει στο κείμενο και γι' αυτό σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει ήδη το κείμενο και αν έχετε και περαιτέρω προτάσεις ευχαρίστω να τις ακούσω και να τις συζητήσω. Αλλά να ξεκινήσουμε με αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν μέσα στο κείμενο και χρειαζόμαστε χρόνο και εσείς για να δείτε το κείμενο και εμείς για να δούμε τις προτάσεις σας και να τις εξετάσουμε επικοδομητικά γιατί νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να επιτύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Γκάλεχερ, μιλήσατε για τα δικαιώματα στην Ιρλανδία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν η Ιρλανδία θέλει μία ρήτρα διασφάλιση για τα δικαιώματα για τον Έθροψ και πει στου ότι μπορείτε να τα πουλήσετε μόνο σε άλλο κάτοχο δικαιωμάτων για το ίδιο ε, είδος, για τον Έθροψ, ε, μπορούν να το κάνουν στην Ιρλανδία. Ναι, μπορούν να τα πουλήσουν σε κάποιον άλλο δικαιούχο για τον έθροπ στην ε, Ιρλανδία. Και βέβαια, γιατί έχουμε πει ότι η πώληση δικαιωμάτων εκτός της χώρας αποκλείεται, απαγορεύεται. Ε, ε, μπορούμε λοιπόν συζητώντας να βρούμε τα ενδεχόμενα κενά και να συμπληρώσουμε αυτά τα οποία χρειάζονται. Τώρα όσον αφορά τις απορρίψεις, η κατάργηση των απορρίψεων δεν είναι εύκολο. Είπαν πολλοί ότι προχωρούμε πολύ γρήγορα, είπαν κάποιοι άλλοι ότι δεν προχωράμε αρκετά γρήγορα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάποια είδη που έχουν μεγάλη εμπορική αξία και να προσπαθήσουμε ε, να θέσουμε ένα τέλος στην απόρριψη για, αυτά, για αυτό το είδος ελίας. Τι θα γίνει λοιπόν, να απαντήσω στην ερώτησή σας, τι θα γίνει αν κάποιος ελίας ε, εξαντλήσει την ε, ποσόστοση για το γάδο, τότε θα πρέπει να σταματήσει την αλία. Θα πρέπει να σταματήσει την αλία εντελώς. Μετά το έτος 2000 τόσο, δεν θυμάμαι για το γάδο πότε ισχύει, ποια χρονιά είναι. Για τα πλέον πολύτιμα είδη λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει για αυτά τα είδη πρώτα απ' όλα η αλία. Δίνουμε λοιπόν ε, κίνητρα για να ακολουθήσουμε μια ε, πιο, πιο επιλεκτικά ε, αλλιευτικά εργαλεία και θα δώσουμε και κίνητρα για την αλλίευση γάδου αν είναι συμβατός ο αλλιέας με, με τους κανόνες. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά, πάντως σε αυτό το τομέα θα προχωρήσουμε βαθμιαία γιατί θέλουμε σε αυτή την απαγόρευση των απορρίψεων να μπουν περισσότερα είδη, μόνο που θα το κάνουμε με σταδιακή προσέγγιση. Ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα διασφαλίσουμε τους αλληλείς για όσα θα συμβούν. αν θα τους δώσουμε επαρκή χρήματα για μηχανισμούς ε, αποθήκευσης, τι θα γίνει με αυτά τα οποία δεν πολλούνται, αν μπορούν να μεταφερθούν σε φτωχότερους. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους. Όσον αφορά τον εξυγχρονισμό του στόλου, η λέξη εξυγχρονισμός ε, μου αρέσει και σας αρέσει και εσάς, πρέπει όμως να συζητήσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τη λέξη εξυγχρονισμός. Αν ε, με τη λέξη εξυγχρονισμός σημαίνει ότι θα δώσουμε χρήματα στους αλληλείς για να ακολουθήσουν μια πιο οικολογική πολιτική και να έχουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμων και να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους, όλα αυτά είναι θετικά. Αυτό εννοούμε όμως ή εννοούμε απλώς αύξηση ε, του δυναμικού του στόλου και των σκαφών. Γιατί στο παρελθόν αυτό γινόταν, αυξάναμε το δυναμικό των σκαφών. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για να μπορέσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε περισσότερα χρήματα για αύξηση της αλλιευτικής ε, ικανότητας. Έχουμε μια πολύ αυστηρή έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο που δεν μας επιτρέπει να δώσουμε χρήματα για τη διάλυση σκαφών από εδώ και πέρα, άρα και αυτή την έκθεση πρέπει να την έχουμε κατά νου και να την τηρήσουμε. Όσον αφορά την ε, συμβατότητα με άλλες πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μια συνεκτική πολιτική και ε, η δίκαιη πολιτική μεταξύ αυτών τα οποία πολλούμε και αυτά τα, αυτών τα οποία καταναλώνουμε δεν είναι εύκολο γιατί αυτό το οποίο κάνουμε εδώ ε, σχετίζεται και με άλλες πολιτικές όπως η πολιτική εμπορίου και άλλες πολιτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν με όλους να συνεργαστούμε και σας διαβεβαιώνω ότι ήδη έχουμε κάνει πολλά βήματα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Αν εσείς όμως έχετε να μου προτείνετε κάτι, πάντοτε τηρώντας τις υποχρεώσεις μας έναντι του ΠΟΕ που όλοι από κοινού έχουμε δεχθεί, εγώ πάντοτε θα είμαι πρόθυμη να σας ακούσω και να συζητήσω τις προτάσεις σας. Όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, Καταλαβαίνω τις ανησυχίες για περιβαλλοντικά και άλλα ζητήματα. Θέλω όμως ε, να είμαι απόλυτα ανοιχτή από αυτού. Πώς μπορούμε να δώσουμε μια εναλλακτική λύση στις ε, χώρες μας έναντι της υπεραλίευσης. Αν δεν δώσουμε τη δυνατότητα σχεδίων υδατοκαλλιέργειας, τι άλλη εναλλακτική έχουν ε, σε σχέση με την υπεραλίευση θα έχουμε μικρότερα, μικρότερες ποσότητες αλίευσης και μεγαλύτερες εισαγωγές από άλλες χώρες που θα έρθουν και θα μας πουλάνε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Και αυτό δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την υδατοκαλλιέργεια και υπάρχει μεγάλο συμφέρον από κράτη-μέλη, όχι μόνο παράκτια κράτη-μέλη, αλλά και κράτη-μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Και εδώ έχουμε και δυνατότητα δημιουργία θέσεων απασχόληση και ανάπτυξη. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραμελήσουμε την ανάγκη για ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας. Το καταλαβαίνω ότι είναι ένα από τα επίμαχα ζητήματα, αλλά και εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση. Όσον αφορά τις ε, απομακρυσμένες περιοχές, θα εξετάσουμε τα αιτήματά σας, πάντοτε έχοντας κατά νου το ισχύον καθεστώς και τη σχετική σταθερότητα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως ε, με αυτό που είπε η κυρία Γόντουστ και ο κύριος Αντινόρο, καθώς και άλλοι ομιλητές, ότι εδώ αυτό που έχουμε είναι ένα έγγραφο εργασίας το οποίο προσφέρετε και μπορείτε πάνω σε αυτό να δουλέψετε. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο δυνατό έγγραφο, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα καλό έγγραφο που μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για την αλλαγή που θέλουμε να επιφέρουμε. Αναφέρεται σε όλα τα σημαντικά ζητήματα, τίποτα δεν έχει μείνει απ' έξω και ε, ακολουθούμε μία ε, πολιτική ε, με τρόπο δραστήριο και ενεργητικό. Υπάρχει χώρος για τις δικές σας τροπολογίες, υπάρχει και χρόνος για την δική σας συνεισφορά και σα διαβεβαιώ ότι με μεγάλη μου χαρά θα περιμένω τις προτάσεις σας και τις τροπολογίε σας. Αλλά βέβαια πρέπει να καταλάβετε ότι έχετε και πολύ διαφορετικές απόψει μεταξύ σας. Και είναι σαφές αυτό, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή αυτό που θέλει είναι μια ισορροπημένη πρόταση. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα εκ μέρους όλων των συναντέλφων να, ευχαριστήσω την Επίτροπο η οποία ήρθε στην Επιτροπή μας σήμερα για να μας ε, παρουσιάσει τη δέσμη των μεταρρυθμίσεων. Να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα το ότι είστε ανοιχτοί στο διάλογο. Ο Πολωνός Υπουργό και Προεδρεύου του Συμβουλίου σήμερα το πρωί μας πρόσφερε συνεχή διάλογο για το τόσο σημαντικό αυτό τομέα και θέμα και σα εγγυώμαι και εγώ από πλευρά μου ότι θα διατυπώσουμε ω κοινοβουλίου συνενετικέ προτάσεις και δεν θα δώσουμε όλες μας τις εξουσίες στα γνωμοδοτικά ε, συμβούλια. Ίσως ε, προχωρήσουμε με έναν ενδιάμεσο τρόπο, προσπαθώντας να καταλήξουμε σε κάποιο συμβεβασμό και ίσως και να βελτιώσουμε τις δικές σας προτάσεις. Σας ευχαριστούμε. Εμείς θα αρχίσουμε σοβαρά τώρα να επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό Ah, bueno, no, pero voy a la Gracias eh, por todo. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Λοιπόν, θα έχουμε συνάντηση των συντονιστών, αλλά πριν από αυτό να πω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας θα είναι την 31η Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30.